Uh, Το επόμενο θέμα ε, είναι η ε, σύσταση της ε, κυρίας Γκροστέτ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνορικής υγειονομικής περίθαλψης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα λάβω τον λόγο για τέσσερα λεπτά και θα κρατήσω τα δύο άλλα λεπτά για το τέλος της ζήτησης. Κύριε Πρόεδρε, κυρία μάλλον, εκπρόσωπο του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, θα έλεγα ότι βλέπουμε την άκρη της σύραγγας για αυτό το σημαντικότατο θέμα για τους ασθενείς. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε με αυτήν την ασαφή κατάσταση όπου ε, το δίκαιο ήταν αυτό της Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχουμε τώρα σαφείς κανόνες για την κινητικότητα και την κυκλοφορία των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι περίθαλψη μπορεί κανείς να έχει στο εξωτερικό, με βάση ποια κριτήρια μπορεί κανείς ε, να λάβει επιστροφή των δαπανών. Πώς γίνεται ε, με την χώρα από την οποία τη σχέση ανάμεσα στην χώρα προέλευσης και στην χώρα που περιθάλπεται. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Βελγική ε, Προεδρία για την εξαίρετη εργασία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, την ικανότητα πειθούσα που ήταν αποφασιστική, διότι πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν επιθυμούσαν αυτή την οδηγία και νομίζω ότι επρόκειτο για ανευθυνότητα. Θα ήθελα επίσης να αποτίσω φόρο τιμής σε φίλο ε, και παλιόν βουλευτή John Bowies που βρίσκεται στα θεωρία πως εισηγητής πρώτης ανάγνωσης και αυτός ήταν ε, δημιουργός αυτής της οδηγίας και ε, πάντοτε συνηγορούσε υπέρ των δικαιωμάτων των ασθενών. Ευχαριστώ επίσης τον Επίτροπο Νταλή και τους συναδέλφους όδες συζητητές που συνέβαλαν, συνέβαλαν ενεργά στην κατάληξη των διαπραγματεύσεων, διότι χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε καταστεί εφικτό. Ποιο είναι εδώ το διακύβευμα για τους ασθενείς. Ε, το, λόγω προόδου ιατρικής ε, η προσφορά δεν μπορεί να είναι προσφορά ε, καθαρά εθνική για όλα τα νοσήματα και κανείς θα πρέπει ε, να διασχίσει τα σύνορα για μια περίθαλψη. Αυτό ε, ισχύει για άτομα που ζουν δίπλα στα σύνορα ή διότι υπάρχουν περισσότερα μέσα και γνώσεις σε ένα άλλο κράτος μέλος, όπως για μερικές εξειδικευμένες θεραπείες και για μερικούς Ευρωπαίους είναι πιο πρακτικό να λάβει κανείς ε, περίθαλψη εκτός της χώρας του, διότι έχουν συγγενείς που ζουν σε άλλη χώρα μέλος. Οι καταναλωτές, οι μισθωτοί, οι και ε, τώρα οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν το δικαίωμα κινητικότητας μέσα στην Ένωση χάρη σε σαφείς νομοθετικές διατάξεις. Ε, βεβαίως ε, δεν πρόκειται να ενθαρρύνουμε ιατρικό τουρισμό, διότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και η διαχείρισή τους είναι της πλήρους αρμοδιότητας των κρατών μελών. Οι ασθενείς θα μπορούν εφεξής σε ένα άλλο κράτος μέλος να λάβουν όλη την περίθαψη που δικαιούνται ε, στην χώρα τους ε, και να τους επιστραφούν οι δαπάνες ε, για ε, όπως και στη χώρα τους για τις, ε, την νοσοκομιακή περίθαλψη με μία διανυκτέρευση ή για δαπανηρές θεραπείες θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης. Υπάρχει λοιπόν μια αναγκαιότητα προγραμματισμού και επενδύσεων των κρατών μελών στο σύστημα περίθαλψής τους. Ε, οι όροι άρνησης θα πρέπει να είναι περιορισμένοι και να υπάρχουν σε έναν κατάλογο κλειστό ε, Λόγω της ασφάλειας των ασθενών επίσης πετύχαμε άλλες πρόοδους. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει, να δημιουργήσει σημεία επαφής εθνικά για να προσανατολίζει καλύτερα ε, τον ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Κάθε σημείο θα είναι μια μοναδική θηρίδα, ένα one-stop shop και ο ασθενής θα έχει έτσι σαφής και ακριβής πληροφορία. Στο θέμα της επιστροφής των δαπανών που ήταν σημαντικό εμπόδιο, έχει βελτιωθεί εκεί η κατάσταση, θα μπορεί κανείς είτε να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης όπως ε, με την Οδηγία Κοινωνικής Ασφάλισης 883 του 2004 ή θα μπορέσει να προκαταβάλει τις δαπάνες ο ασθενή και να λάβει επιστροφή το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες να μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν μια γνωμοδότηση στο εξωτερικό για διάγνωση της ασθένειας και για να δοθεί άδεια για περίθαλψη. Και κλείνω λέγοντας ότι χάρη στην ευρωπαϊκή συνεργασία σε τομείς όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς οι ασθενείς έτσι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολύ εξειδικευμένη ε, περίθαλψη και έτσι αυτό ενθαρρύνεται, κανεί, ενθαρρύνεται ε, το μοίρασμα, η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και διαγνώσεων. Έτσι νομίζω ότι φτάσαμε στο στόχο μας και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και μπορώ να πω ότι έτσι η Ευρώπη της υγείας οικοδομείται διαμέσου της οδηγίας αυτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιώρη, εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κυρία Γκροστέτ, ε, αγαπητά μέλη του σώματος, θα συνεχίσω στα Ουγγρικά. Χαίρομαι διότι είμαι σε θέση να συζητήσω τα δικαιώματα των ασθενών μέσα στα πλαίσια των, της διασυνοριακής περίθαλψης. Διανύουμε ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, διότι μετά από δύο χρόνια εκπόνησης φτάνουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν αυτή τη διαδικασία. Τα δύο προγενέστερα μέλη την Ισπανία και το Βέλγιο για την εξαιρετική εργασία που επιτέλεσαν τα δύο άλλα μέλη της Τρόικας για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό στο Συμβούλιο. Εξ του Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία και την ετοιμότητα για συμβασμό. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει τους ασθενείς παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ασθενών στην Ευρώπη. Οι συζητήσεις δεν ήταν εύκολες, αλλά πάντα ήταν επικοδομητικές και προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ξέρω ο, ότι και εσωτερικές σας διεργασίες ήταν καθόλου εύκολες και η έκθεση που θα ψηφίσετε αύριο είναι απότοκη ενός συμβιβασμού μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό το συμβιβασμό. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκροστέτ προσωπικά, καθώς και όλους τους σκιώδεις, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατόν να επιτύχουμε σε αυτό το νομοθετικό σχέδιο. Είμαι σίγουρη ότι η νέα αυτή νομοθετική βάση θα οδηγεί σε μια εξισορρόπηση μεταξύ δικαιωμάτων των ασθενών και των υποχρεώσεων των κρατών μελών να οργανώσουν την υγειονομική περίθαλψη μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους. Καταφέραμε να φτάσουμε σε αποδεκτές λύσεις για μια σειρά προβλημάτων και ζήτημάτων. Καταρχήν, καταφέραμε να εξεύρουμε μία λύση σε σχέση με την ε, ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και βρήκαμε μία λύση ως προς το σύστημα προέγκρισης και επιστροφής εξόδων για τις δαπάνες στη διασυνοριακή περίθαλψη. Επίσης, φτάσαμε σε μία συμφωνία για τους ασθενείς που πάσχουν από μία σπάνια ασθένεια. Και επίσης, θα δούμε και θέματα ε, ηλεκτρονικής περίθαλψης, e-health. Νομίζω ότι φτάσαμε σε μία πολύ καλή συνεργασία Επιτύχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και ε, φτάσαμε σε μια συμφωνία που σέβεται και τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς διασυνοριακά και θα ήθελα να τονίσω και τη σημασία των εθνικών σημείων επαφής. Η αμοιβαία αποδοχή συνταγογράφησης είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ο κανονισμός 883 κάθετος 2004 για τον συντονισμό ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει οδηγήσει σε ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια των ασθενών. Τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από αρχές που έχουν αναφερθεί από όλα τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή μιλάμε για ισοτιμία και αλληλεγγύη. Και επίσης βρήκαμε ορισμένες ατραπούς για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την ε, λειτουργία των συστημάτων υγείας. Η Ουγγρική Προεδρία έχει αναλάβει τη δέσμευση να περάσει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Παραμένουν θέματα καθαρά συντακτικά και όταν διευθετηθούν θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κινητήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Ντάλι, εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μεγάλο επίτευγμα ε, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για την οδηγία αυτή. Είμαι δίδρα ευγνώμων προς τον εισηγητή, προς την ε, εισηγητρία μάλλον, την κυρία Γκροστέτ, τους κοιόντους εισηγητές για τη σκληρή τους δουλειά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ασθενών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανία και το Βέλγιο τις δύο προηγούμενες προεδρίες για τη δουλειά που έκαναν για να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος. Νομίζω ότι η νέα οδηγία θα αποτελέσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Επίσης θα δημιουργήσει μια νέα φάση συνεργασίας, αν θέλετε, μεταξύ των 27 εθνικών συστημάτων υγείας δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί η σημερινή συμφωνία. Θυμάμαι πέρσι όταν ήρθα, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μου είπαν πολλοί ότι οι διαπραγματεύσει για την οδηγία είχαν φτάσει σε αδιέξοδο. Η οδηγία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για την ανάγκη πολιτικής ηγεσία και καταδεικνύει ότι με αποφασιστικότητα και θάρρος μπορούν να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις προς όφελος των πολιτών μας. Θεωρώ ότι τα νομοθετικά όργανα δεν πρέπει να αφήνουν το δικαστήριο να αποφαίνεται ε, αντί για αυτά. Είναι πιο σωστό να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ασθενών παρά να χρειάζεται να πηγαίνουν στο δικαστήριο. Αναγνωρίζεται λοιπόν ο λόγος, ο ρόλος του νομοθέτη να εξασφαλίζει τα δικαιώματα αυτά. Να σας αναφέρω κάποιες από τις απόψεις που αναφέρονται στην οδηγία. Καταρχάς, είναι σαφές ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν καθήκον να επενδύουν στο εθνικό του σύστημα για να προσφέρουν στους πολίτες τους χωρίς καθυστέρηση την φροντίδα που χρειάζονται. Έτσι λοιπόν η οδηγία θα συμβάλλει στη μείωση ε, των προβλημάτων των εμποδίων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι ασθενείς θα μπορούν να δουν τον ε, περιθάλποντα της επιλογής τους ε, όποτε θέλουν. Όταν ο χρόνος αναμονής όμως είναι υπερβολικά ε, μακρύς, ο ασθενής θα μπορεί να αποτανθεί σε άλλο κράτος μέλος και να τα επιστραφούν τα έξοδα. Ωστόσο, τι ορίζουμε ως καθυστέρηση. Αυτό θα πρέπει να το ορίσουμε με προσοχή. Η βασική πρόοδος που επιτυγχάνεται με την οδηγία αυτή σε σχέση με την τρέχουσα νομοθεσία είναι ότι οι ασθενείς θα έχουν την επιλογή να πρόσβαση μάλλον στον θεράπονται οι ιατρό της επιλογή τους για να ε, τους εγγυάται η ποιότητα της περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, η οδηγία θα δώσει στους ασθενείς πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά τους και την διασυνοριακή περίθαλψη. Ε, αυτές τις πληροφορίες θα τις δίνουν τα, κέντρα, εθνικά κέντρα ενημέρωσης, όχι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Και τρίτον, αναφέρεται η οδηγία στην ποιότητα της περίθαλψης. Δίνεται διαφάνεια σε σχέση με τα εθνικά πρότυπα. Θα υπάρξει λοιπόν μια σύγκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ποιότητα της περίθαλψης. Και τέλος, η οδηγία θέτει τη βάση για ευρωπαϊκή συνεργασία σε ό,τι αφορά την υγεία. Είναι μεν τελούσια τα δίκτυα τα οποία δημιουργούνται από την οδηγία, αλλά είμαι βέβαιος ότι τα κάτι μέλη θα διαπιστώσουν ότι πολλά έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία τους. Είναι θέμα αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν βασίζομαι στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία και ούτω καθεξής. Επίσης η οδηγία προβλέπει ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς για την ε, ενημέρωση σε σχέση με την τεχνογνωσία για θέματα υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρε, ε, Υπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, η τελική, ο τελικός συμβιβασμός που έχουμε μπροστά μας σήμερα αποτυπώνει το πνεύμα της ε, οδηγίας για τη βελτίωση της διασυνοριακής περίθαλψης λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Είναι μια καλή ημέρα για την Ευρώπη της υγείας. Τέλος, να κάνω την εξής δήλωση για ένα θεσμικό στοιχείο του κειμένου. Έχει η Επιτροπή της αμφιβολίες της κατά πόσον κάποια στοιχεία θα εφαρμοστούν ως εφαρμοστικές πράξεις. Όταν ε, ασκεί τις εφαρμοστικές της αρμοδιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα χρησιμοποιήσει της κατεξουσιοδότηση πράξης βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λίζε έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπε, Υπουργέ, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι σημαντική ημέρα για τους ασθενείς στην Ευρώπη, όντως, γιατί ήταν ε, απαράδεκτο να έχουμε το δικαίωμα να πάμε σε ένα άλλο ε, κράτος μέλος, το οποίο το έχει αναγνωρίσει και το ΔΕΚ, αλλά πολλά κράτη-μέλη δεν το είχαν ε, εφαρμόσει αυτό. Και σε κάθε ασθενή του έλεγαν να πάει στα δικαστήρια μέχρι ότου να καταλήξει στο ΔΕΚ σε πολλές περιπτώσεις. Θεωρώ ότι είναι κοινική αυτή η αντιμετώπιση και είναι, ε, ξέρετε, αδύναμοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άρρωστοι, αλλιώς δεν θα χρειάζονταν περίθαλψη και στην τελική ανάλυση μπορεί να έχουν πεθάνει μέχρι ότου να αποφανθεί το ΔΕΚ. Γι' αυτό λοιπόν είναι καιρός να δημιουργηθεί σαφήνεια, νομική σαφήνεια και για τους ε, ασθενείς που εφαρμόζονταν λίγο πολύ τα ζητήματα αυτά πετύχαμε πολλά, πολλές επιτυχίες όπως τα εθνικά σημεία επαφής, τα δίκτυα αναφοράς και εδώ υπάρχει λοιπόν βελτίωση σε σχέση με τις χώρες εκείνες όπου λίγο πολύ εφαρμόζονταν οι αποφάσεις του 10 για μια Ευρώπη της υγείας, όπως είπε και ο Επίτροπος. Δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να αφιερώσω τα 15 τελευταία δευτερόλεπτα για να, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ντάλη και τον Τζον Μπόις, κυρίως ο οποίος είναι εδώ πέρα στα έδρανα πάνω, ο οποίος είναι ιδρυτής αυτής της οδηγίας. Τον ευχαριστώ πολύ και τον συγχαίρω. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ροτμπέρεντ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είναι περιττή αυτή η νομοθεσία ουσιαστικά και ελπίζω να, είναι, να παραμείνει περιττή νομοθεσία γιατί δεν θα χρειαστεί να την εφαρμόσουν, να τη χρησιμοποιήσουν οι ασθενεί. Γιατί στην ιδανική περίπτωση, στον ιδανικό κόσμο, οι ασθενεί θα πρέπει να έχουν την περίθαλψη στην χώρα η οποία, στην οποία ζουν, στην οποία έχουν γεννηθεί ίσω και το γεγονός ότι πρέπει να συζητήσουμε, συζητάμε τα πράγματα αυτά εδώ είναι κοινικό. Έχετε δίκιο. Γιατί αυτή σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει αυτό που οφείλουν στους πολίτες τους, δηλαδή γρήγορη ποιοτική ε, περίθαλψη, υγειονομική περίθαλψη και καταδεικνύει ότι προτιμούν να επενδύουν σε άλλους τομείς και όχι σε αυτόν τον τομέα για τους πολίτες. Είναι ντροπή. και αν αυτή η οδηγία κάποια στιγμή εφαρμογή, εφαρμοστεί, αν τη χρειαστούν οι ασθενείς, θα είμαι ευτυχισμένη, ευτυχής που πετύχαμε αυτά που πετύχαμε και ευχαριστώ την κυρία Γκροστέτ για αυτά που πετύχαμε. Πολλά πετύχαμε. Πετύχαμε επιτέλους οι σπάνιες ασθένειες να τεθούν στο επίκεντρο της προσοχής μας, γιατί πάντα αυτοί που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες ήταν ε, στο περιθώριο. Επίσης, ε, επιτέλους καταφέραμε άνθρωποι να έχουν σημεία επικοινωνίας, ενημέρωση στα κράτη-μέλη να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους. Δεν υπήρχε αυτό ω τώρα. Και αν στο μέλλον δημιουργηθούν δίκτυα αναφοράς θα υπάρξει επιτέλους ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν υπάρχει σε συντονισμένο επίπεδο. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, αλλά όχι έτσι συντονισμένα. Όλα αυτά είναι τεράστια επιτεύγματα χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Φυσικά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία με δυσαρεστούν. Αυτό το θέατρο, αυτή η διαφωνία για την πρώτερη έγκριση θα ήθελα να είχαν διαμορφωθεί διαφορετικά τα πράγματα γιατί αυτό θα έδειχνε ότι είναι πιο σοβαρά τα κρατημέλη. Ο στόχος ωστόσο, συνάδελφοι, θα πρέπει να είναι το υγειονομικό σύστημα περίθαλψης να είναι τόσο καλό σε κάθε κράτος μέλος που κανείς να μην θέλει να φύγει σε άλλη χώρα. Και αν κάναμε ένα μικρό βήμα σήμερα και γιατί δημιουργήσαμε διαφάνεια, πετύχαμε πολλά. Ελπίζω να είναι, λοιπόν, να υπάρξει αυτή η συνέπεια σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Προέρχομαι από ένα κρατος μέλος όπου τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα, αλλά ξέρω ότι σε άλλες ε, χώρες ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και γι' αυτό ντρέπομαι, γιατί είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα αυτή. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ όμως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ντάλη και την ομάδα του και τον ε, πατέρα της, του συμβιβασμού αυτού του κυρίου Μπόης να ευχαριστήσω και τη Βελγική Προεδρία που έκανε ό,τι μπορούσε για να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Και ήταν πράγματι πάρα πολλά αυτά που έκανε η Βελγική Προεδρία, αν κοιτάξουμε και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες δεν κινούνται καθόλου προς τα εμπρός. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εξετάζοντας πριν τέσσερα χρόνια, όταν είχαμε την εκστρατεία για τους ασθενείς, ε, χαιρέτησα την ε, συμφωνία το Δεκέμβριο. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Γκοστέτ και τους κοιόδης εισηγητές για την καλή συνεργασία και ξέρετε εργασία που επιτελέστηκε όπως επίσης και το δημιουργό ε, Μόρις αυτής της πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ Τζον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, ήταν ενωμένο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Υποστηρίξαμε τους ασθενείς και θα υπάρξει σαφώς ένα πλαίσιο νομοθετικό σαφές για περίθαλψη σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η συμφωνία είναι ένα μικρό βήμα, αλλά είναι πρόοδος για τους ασθενείς που θα ενισχύσουν τα δικαιώματά τους ε, και θα έχουν καλύτερες γνώσεις και καλύτερη ποιότητα περίθαλψης. Βεβαίω θα είχαμε υποστηρίξει κάτι το πιο φιλόδοξο, παρόλο που είναι ανάγκη τα κράτη-μέλη ε, να έχουν προγενέστερη ε, αδειοδότηση για το θέμα αυτό. Βεβαίως η Βελγική ε, Προεδρία βεβαίως ε, έχει ε, δώσει περισσότερη σημασία σε οργανωτικά θέματα από την ίδια την περίθαλψη. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Η ποιότητα και η ασφάλεια ως ε, κριτήριο για απόρριψη των προτεραιοτήτων τα κράτη-μέλη ήταν αντίθετα για κάθε σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και αναβάθμισης ε, της ε, περίθαλψης. Χαιρετίζω την μελλοντική οδηγία αλλά θα είμαστε αυστηροί για την εφαρμογή και θα πρέπει να υπάρξει εποπτεία, παρακολούθηση, αναφορές και εκθέσεις για να δούμε αν εφαρμόζεται καλά η οδηγία και να μην υπάρχουν εμπόδια για τους ασθενείς. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχει έλλειψη φιλοδοξίας για την συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρονικής ε, υγείας. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής έχει ε, στραγγαλιστεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Ντάλη, ε, θεωρείται η Επιτροπή ότι ε, μια πρόταση για την ηλεκτρονική υγεία που θα, προωθεί την ε, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Λάμπερτ, 1,5 λεπτό. Πολλοί εδώ θα θυμούνται ότι στην πρώτη ανάγνωση πρόκειται για ένα πολύ φλέγον ζήτημα και ακούμε μερικές από τις διαφωνίες ανάμεσά μας. Υπήρξαν ανησυχία αν οι ε, δυνάμεις ε, της αγοράς θα υπερίσχυαν του δημοσίου συμφέροντας ε, και του δικαιώματος των ασθενών να επιλέγουν και να ταξιδεύουν. Μερικοί λέγανε ποιοι είναι οι ασθενείς που θα το επιλέξουν αυτό. Αυτό που έχουμε τώρα τελικά είναι ένας λογικός συμβιβασμός. Όπως λέχθηκε ήδη, για αυτούς που είναι αναγκαίο να έχουν μια κατεπίγουσα περίθαλψη έχουμε ήδη ένα σύστημα συντονισμένο. Αυτή η οδηγία αναφέρεται περισσότερο ε, στην επιλογή, στην ικανότητα των ατόμων να επιλέξουν πού θα πάνε ε, και να τους ακολουθούν ε, και τα κονδύλια. Έχουμε τώρα ε, συστήματα που θα μπορούν να εξασφαλίσουν την κάλυψη αυτών των αναγκών. Η οδηγία αυτή πρέπει να επικροτηθεί διότι αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την νομική διάσταση, την νομική βεβαιότητα για να δούμε ποια θα είναι, που θα, ποιος θα είναι υπεύθυνο για την συνέχεια ε, της ε, ε, θεραπείας, για αποζημιώσεις αν κάτι δεν πάει καλά, για τα προσόντα του ιατρικού επαγγέλματος. Έχουμε επίσης μια καλό συμβιβασμό για τις σπάνιες ασθένειες, πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι στην πρώτη ανάγνωση. Νομίζουμε ότι για πολλούς ασθενείς τα πράγματα θα πάνε καλά, αλλά θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε για τους ασθενείς Στι μας στις δικές μας χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαπανόκ, 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι Πρόεδρε, Επίτροπε, Υπουργέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπόους και την κυρία Γκροστέτ. Έχουν περάσει δύο χρόνια και έξι μήνες από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την, την πρότασή της για την για διασυνοριακή περίθαλψη, αλλά οι σχετικές εργασίες είχαν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Αυτό το θέμα ήταν μέρος της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες και κάναμε λοιπόν το λάθος να εξαιρέσουμε τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η οδηγία αυτή, η τρέχουσα, αναφέρεται μόνο σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, τα συστήματα κοινωνικής, μάλλον υγειονομικής περίθαλψης βασίζονται σε κοινέ αρχές, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο διοργανώνονται σε κάθε κράτος μέλος. Η πρόταση που θα ψηφίσουμε σήμερα και την οποία θα υποστηρίξω είναι, ε, αποτελεί ένα συμβιβασμό μεταξύ των ε, δικαιωμάτων των πολιτών και των ασθενών αφενός και των ε, φόβων των κρατών μελών αφετέρου. Η σημερινή πρόταση αποτελεί ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα προς τα μπροστά. Το σχέδιο οδηγίας ε, ξεκαθαρίζει τα δικαιώματα των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη και στην ενημέρωση, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών για την διοργάνωση και τη χρηματοδότηση των συστημάτων περίθαλψης ορίζεται με και ορίζονται επίσης οι κανόνες για την πρώτερη έγκριση για την ε, νοσηλεία. Ελπίζω κυρίες και κύριοι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω την οδηγία αυτή στα επόμενα έτη και να βελτιώνουμε τα δικαιώματα των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Λίωταρτ. δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν είναι η ώρα της αλήθειας. Η περίθαλψη θα γίνει ένα προϊόν της εσωτερικής αγοράς, ένα εμπόρευμα Όποιος έχει τα πιο πολλά χρήματα θα είναι αυτός ο οποίος θα λαμβάνει την καλύτερη περιθάλψη. Η πρόταση ε, διαιωνίζει αυτό το διχασμό στην περίθαλψη. Αναρωτιέμαι πώς το δέχονται αυτό πολλοί συνάδελφοι. Η περίθαλψη είναι μια βασική ανάγκη που θα πρέπει να έχουν, στην οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι θεωρούν ε, όσοι είναι υπέρ της οδηγίας ότι κάνουν χάρη στους ασθενείς. Αλλά εγώ διαφωνώ, εγώ είμαι υπέρ όσων ωφελούν τους ασθενείς. Αλλά πολλά ε, είναι τα στραβά εδώ της οδηγίας. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Οι ασφαλιστές θα θέλουν να στέλνουν τους ε, ασθενείς για διασυνοριακή περίθαλψη, αν είναι πιο φτηνή αυτή αλλού. Η περίθαλψη η η οποία δεν είναι πλέον αποδοτική οικονομικά θα εξαφανιστεί από τις πιο α, πλούσιες περιοχές. Δεν πρόκειται για δικαιώματα αλλά για υποχρεώσεις των ασθενών. Οι ασθενείς σε πιο φτηνές περιοχές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε άλλη περιοχή γιατί τα επιπλέον έξοδα δεν θα επιστρέφονται αυτόματα. Άρα ο τουρισμός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα ωφελήσει τους ε, πιο ευκατάστατους. Οι περιοχές δε με μικρές ε, λίστες αναμονής θα, θα φτάσουν να έχουν τόσο πολλούς ε, τουρίστες στον τομέα της περίθαλψης που δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αναφέρονται σχετικά ζητήματα και στη βελγική εφημερίδα The Standard και να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα παραδείγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περίθαλψη για τους ασθενείς όσο πιο κοντά γίνεται στη δική τους γλώσσα, κοντά στην οικογένειά τους. Και αντί να φροντίσουμε γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει την αγορά να δουλέψει. όποιο συμφωνεί με αυτό θα υπερψηφίσει αύριο την οδηγία. Όποιος συμφωνεί μαζί μου θα την καταψηφίσει σίγουρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση, ένα μισή λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν η οδηγία είχε ορισμένα κρίσιμα σημεία. Ο τριμερής διάλογος οδήγησε σε ένα εξισορροπημένο κείμενο που λαμβάνει υπόψη τις ποιοτικέ απαιτήσεις της υγειονομικής περίθαλψης, στην αρχή της επιστροφής εξόδων, της προέγκρισης και την ε, αντιμετώπιση σπανίων νόσων. Θέλουμε να έχουν όλοι οι ασθενείς δικαίωμα στην ε, υγειονομική περίθαλψη εκτός συνόρων, χωρίς να προωθήσουμε τον ε, ιατρικό τουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν η χώρα προέλευσης να αναλαμβάνει τα έξοδα. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν υψηλά επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης αλλά αυτό δεν στάθηκε δυνατόν. Επειδή θέλουμε να ταχθούμε υπέρ του, της έκβασης της συζήτησης, θα υπερψηφίσουμε. Όπως θα ισχύσει και για την εντόπιση του Αλσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενοποίηση των ε, υπαρχουσών πολιτικών. Θα θέλαμε να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών υπέρ των ίδιων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζεκέντη. Ζεκέντη για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, είμαι υπέρ της διασυνοριακής περίθαλψης και των δικαιωμάτων των ασθενών. Διάφορα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς επιζητούν, επιδιώκουν διασυνοριακά περίθαλψη και γνωρίζουμε την περίπτωση του Λουξεμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη ανατολικά και ε, δυτικά και αυτές ε, οι διαφορές ε, είναι ακόμα μεγαλύτερες από απλά διαφορές οικονομικές, είναι διαφορές της ευκαιρίες επίσης. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να μειώσει αυτές τις διαφορές και το χάσμα. Αν έχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε όλα τα κράτη-μέλη θα μειώσουμε την ανάγκη που αισθάνονται οι ασθενείς να πηγαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη για περίθαλψη. Εκτός τούτων, πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να συντονίσουμε τις ιατρικές απόψεις περιθεραπείας για διάφορες ασθένειες, διότι η υγεία είναι κάτι το οποίο όλοι δικαιούνται και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ε, ε, να υπάρχει μεταχείριση διαφορετική για έναν Ούγγρο από ό,τι για έναν Σουηδό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλνερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες τις οποίες έχω ζήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο γιατί αφορά τόσο πολλά άτομα. Οι πιο πολλοί Άλλωστε θέλουν να έχουν ε, πρόσβαση στην περίθαλψη εκεί που ζουν. Αλλά μιλάμε για θέματα ζωής ή θανάτου σε πολλές περιπτώσεις και αυτή είναι η βασική σκέψη πίσω από την ευρωπαϊκή συνεργασία. Το θέμα είναι να διευρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία για αυτούς που τη χρειάζονται πιο πολύ από κάθε άλλον, για τους ασθενείς, τους ε, αρρώστους. Πρόκειται σίγουρα για ένα συμβιβασμό και ξέρω και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι, ότι το ΕΛΚ θα ήθελα να έχει προχωρήσει περαιτέρω σε πολλά ζητήματα, αλλά... Όταν μας μιλάνε για τουρισμό υγείας, για κατάρρευση των συστημάτων υγείας, πρέπει να σας απαντήσω ότι δυστυχώς υπάρχει το θέμα αυτό με την πρώτερη έγκριση ε, όταν θέλει κανείς να πετύχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά που έχουμε πετύχει, τα έχουμε πετύχει παρά τη Σουηδική Αριστερά, όχι σε συνεργασία με τη Σουηδική Αριστερά, να σας το πω έτσι, χτες αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το, το σύστημα της πρώτης έγκρασης και στην Σουηδία. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Αυτό εξαρτάται όμως πλέον από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε καλύτερη περιθάλψη, όχι να την περιορίσουμε. Αυτή είναι η κλίση που απευθύνει λοιπόν και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προσέξει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Παρνιό. Euh, Madame la Présidente, tout d'abord, permettez-moi euh, d'affirmer notre satisfaction face aux progrès mis en œuvre par cette directive que nous allons voter demain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 Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ε, αυτό, αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της διασυνοριακής περίθαλψης. Εάν ε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα διασυνοριακού τουρισμού, αλλά θα πρέπει να θεωρήσουμε την υγεία όχι ως ε, ένα εμπόρευμα. Μιλάμε για ίσα δικαιώματα. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια μιλήσαμε για την αρχή προέγκρισης, ιδιαίτερα για την νοσοκομιακή περίθαλψη και την περίθαλψη εκτός νοσοκομείου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ε, Γκροστέτ και την κυρία Ροτ Μπέρεντ γιατί προωθήσαμε το όλο ζήτημα μέσα στα πλαίσια της ε, επιστροφής εξόδων και ενός ευρωπαϊκού δικτύου αναφοράς αντιμετώπιση των σπανίων νόσων και ε, συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Δεν έχει λήξει όμως η εργασία μας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω έτσι ώστε να διαγράψουμε τις διαφορές που υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε αυτή η ίση μεταχείριση να συνεχίσει να υφίσταται και για τον ασθενή αλλά και για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λεπάζ, για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, Καταρχήν αυτή η συμφωνία διασαφηνίζει από νομικής πλευράς το ζήτημα διότι μέχρι τώρα αποφαινόταν το ΔΕΚ, δηλαδή υπήρχε ανασφάλεια δικαίου. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς την κυρία Γκροστέ, του Σκιώδης, καθώς και την εργασία του Επιτρόπου Νταλή. Έτσι υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση των ασθενών καθώς και ποιότητα παροχής υπηρεσιών και μείωση του κόστους. Είμαι υπέρ του συστήματος προέγκρισης για τις πιο βαριές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα ο ασθενής να δεχτεί την περίθαλψη στο εξωτερικό, στην Αλοδαπή, μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Όμως ως προς τους όρους εφαρμογής αυτής της οδηγίας νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ανισότητα μεταχείρισης μεταξύ ασθανών. Τι σημαίνει εύλογη προθεσμία θα πρέπει αυτή η εύλογη να μην ε, διακυβεύσει τα δικαιώματα των ασθενών. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ορίσουν χρηματοδοτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε οι φτωχότεροι ασθενείς να μην επομίζονται πολλά έξοδα. Δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε ε, την ύπαρξη διοικητικών προσκομμάτων που να συρρυκνώσουν τα δικαιώματα του ασθενούς. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν ανισότητες ως προς την επιστροφή εξόδων, εάν υπάρχει ελάχιστη ε, επιστροφή ή μεγαλύτερη σε άλλες περιπτώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να προβάλλω. Ο κύριος Τούρμες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Τζον, η οδηγία αυτή δημιουργεί ε, σαφή και διαφανή δικαιώματο και έτσι η στάση στο εξωτερικό είναι πλέον ε, σαφής και όχι αυθαίρετη όπως ήταν σε κάποια κράτη-μέλη. Η οδηγία αυτή θα οδηγήσει σε καλύτερη πληροφόρηση για την περίθαλψη στο εξωτερικό. Ωστόσο, η οδηγία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί κιόλα από τις κυβερνήσεις. Αυτό που η οδηγία αυτή ωστόσο εμποδίζει είναι αυτό που κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ονειρεύονταν και ίσως και εδώ. Δηλαδή να ανοίξουν οι σε σύνορα προκειμένου να βελτιωθούν τα εθνικά συστήματα υγείας και είμαι περήφανος που με τους δύο εισηγητές καταφέραμε να τηρήσουμε τις ισορροπίες αυτές. Να πούμε όχι στον ε, ε, τουρισμό της υγείας, ε, και να διατηρηθούν τα εθνικά συστήματα. Οι ποιοτικέ ε, διαφορέ ε, στην ιατροφαρμακευτική περιθάλψη δεν μπορούν να λυθούν με την οδηγία αυτή, αλλά μόνο με επαρκή επενδύσει από τα εθνικά κράτη. Και εγώ θα ήθελα, κύριε Ντάλη, μετά την οδηγία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει πιο πολύ το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας που αποτελεί το θέμα βάσης, να είναι σαφές ποιος πληρώνει τι, να ασκηθεί πιο πολύ πίεση στα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί αυτό παρά να αναπτυχθούν νέες ιδέες ε, απελευθέρωσης και ανταγωνισμού. Ευχαριστώ κύριε Σουίνμπερν. Ευχαριστώ. Αυτή η οδηγία λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ε, για την παγίωση και ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η εφαρμογή θα έχει στην Ουαλία, την εκλογική μου περιφέρεια, μεγάλο αντίκτυπο. Νομίζω ότι η διαχείριση βεβαίως των υγειονομικών υπηρεσιών ανήκει στην κυβέρνηση πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο σχετικά με την ε, κάλυψη, την επιστροφή των εξόδων. Υπάρχει ένα μέτρο ευελιξίας ε, σε αυτές τις προτάσεις, η ικανότητα για τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν για επιλέξιμη θεραπεία με προηγούμενη αδειοδότηση ε, και για την θέσπιση ενός συστήματος επιστροφής των εξόδων θα ελαφρύνει την επιβάρυνση Νομίζω ότι το έργο των συναδέλφων κυρίως του κυρίου Μπόβης δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη ε, με αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή, να υπάρχει και επίσης αναβάθμιση του επίπεδου των υπηρεσιών τους ώστε να είναι καλή η επιλογή των ασθενών. Κύριος Φερέρα. Πρόθεση αυτής οδηγίας είναι απόλυτα σαφής εδώ μιλάμε για απελευθέρωση των υπηρεσιών περίθαλψης έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα, τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς ιατρικούς ομίλους. Θεωρούμε την υγεία σαν ένα οποιοδήποτε εμπόρευμα και οι ασθενείς δεν γίνονται παρά καταναλωτές. Αυτό επαυξάνει τις ανισότητας μεταξύ πολιτών, ιδιαίτερα εκείνους που δεν μπορούν να προσφύγουν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η έγκριση, ακόμα και με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν, θα σήμαινε μεγάλους κινδύνους, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως την Πορτογαλία, διότι θα είχαμε να κάνουμε με πολύ υψηλό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλει ε, υποχρεώσεις δημοσιονομικές, θέλει στην ουσία να προωθήσει ιδιωτικά χρηματοοικονομικά συμφέροντα προωθώντας τον ιατρικό τουρισμό. Επειδή μιλάμε για ένα εμπόρευμα, δεν λάβουμε υπόψη την ασφάλεια των χρηστών, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μη νοσοκομιακή υπερίθελψη Δυστυχώς το σύστημα προέγκρισης δεν προβλέπει αυτή τη διαδικασία. Το 2007 είδαμε ότι η οδηγία Μπόλκενστάιν δεν μπόρεσε να περάσει ορισμένα θέματα ως προς την πτυχή υγείας και τώρα πιστεύω ότι δεν θα περάσουν αυτά τα θέματα επίσης. Πασκά. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι ελαφρώς απογοητευμένος με την τοποθέτηση της Επιτροπής για τα διασυνοριακά δικαιώματα των ασθενών. Το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση δεν ενέκρινε πολλές από τις καλές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είχε δημιουργήσει ήδη μια καλή βάση για την τροποποίηση των κανόνων για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών στους ασθενείς προκειμένου οι ασθενείς ε, υπό συγκεκριμένου όρους να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη που χρειάζονται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και γι' αυτό είναι καλό που στην προετοιμασία της έκθεσης στις διάφορες επιτροπές για την δεύτερη ανάγνωση επανήλθε η αρχική φιλοσοφία της ε, θέσης του Κοινοβουλίου και περάσαμε από την έλλειψη ε, διαφάνεια σε μια αξιοπρεπή λύση. Το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο συζητάμε σήμερα βάσει της νομολογίας του ΔΕΚ παρέχει νέες δυνατότητες και νέα ποιότητα στις υπηρεσίες περίθαλψης προς τους ασθενείς μας και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ευχαριστώ. Μετά από μία νομική δεδαλώδη διαδικασία αύριο θα έχουμε μία νομοθετική βάση για τους πολίτες εκείνους οι οποίοι θα πρέπει να αποτανθούν στην αλλοδαπή για να τύχουν περίθαλψης. Αυτό θα σημαίνει ότι οι πλέον πληροφορημένοι ή τυχεροί θα μπορέσουν να καρποθούν αυτού του πλαισίου όπως αναγνωρίζει το ΔΕΚ με βάση τα εθνικά σημεία επαφής δεν θα πρόκειται για ένα ε, βήμα προς το κενό. Πολλές φορές αντιμετωπίστηκαν και γλωσσικά, οικονομικά και γραφειοκρατικά προβλήματα. Ως προς τη διαδικασία περίθαλψης, ίσως ο ασθενής να χρειαστεί να προβεί σε μία προέγκριση. Και αυτό γίνεται για την προστασία των εθνικών συστημάτων υγείας. Πολλές φορές η διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης καλύπτει τα ιατρικά έξοδα, αλλά σε εκούσια βάση. Θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε μία γενικότερη συζήτηση η οποία προβάλλει έναν κοινό παρονομαστή. Δηλαδή να δώσουμε τέλος στο Γολγοθά χιλιάδων ασθενών ανά την Ευρώπη και φαίνεται ότι το καταφέραμε αυτό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κάβενμπακ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Επιτροπέ, καταλαβαίνω ότι η καθήκον της πολιτικής είναι να συμβάλλει στην ε, ε, καλύτερη ποιότητα ζωής και στον, τομέα της υγείας δεν είναι εύκολο το καθήκον αυτό. Καταρχάς είναι χρέος των εθνικών κρατών να φροντίζουν για την καλή πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη ανεξάρτητα από τα εισοδήματα των ασθενών και από τα έσοδα της περιοχής τους. Παρά όλα αυτά όμως, παρά τα συστήματα υγείας υπάρχουν ε, πάντα περιπτώσεις ασθενών όπου οι ασθενείς ε, αναγκάζονται να βγουν στο εξωτερικό ή θέλουν να βγουν στο εξωτερικό για την περιθάλψή τους. Και εδώ η οδηγία αυτή δημιουργεί το νομικό πλαίσιο, τις νομικές δικλίδες, προκειμένου να μην υπάρξει ε, περί γραφειοκρατία και χωρίς μεγάλη ε, χρηματοοικονομική δαπάνη από τους ασθενείς. Θεωρώ ότι η οδηγία αυτή μετά τις μακρές διαπραγματεύσεις αποτελεί μια επιτυχία, παρά το γεγονός ότι στην εφαρμογή της ε, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ελπίζω πολύ να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής και σας ζητώ να εμείνετε σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες σας και τους φιλοδοξίες σας για την ποιότητα της ε, περίθαλψης, γιατί θέλουμε να εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή περίθαλψη με τα καλύτερα δυνατά πρόταπα ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ευχαριστώ. Κυρία Μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Γκροστέτα ε, που συνέχισε την εργασία του πρώην συναδέλφου κ. Μπόης που είναι εδώ παρόν και τον συγχαίρω επίσης και θα ήθελα να τονίσω το σημαντικό ρόλο της Βελγικής Προεδρίας που κατέβαλε τις αναγκαίες προσπάθειες για να καταλήξουμε σε αυτή τη δύσκολο συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο και ορισμένα κράτη-μέλη των οποίων η θέση ήταν κάπως επιφυλακτική. Αυτή η οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη είναι σημαντική παρόλο που αναφέρεται σε 1% ε, των προϋπολογισμών υπολογισμό Υγεία διότι έχει συμβολική σημασία δηλαδή το νόμιμο δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει περίθαλψη στο εξωτερικό και να του επιστρέφονται τα έξοδα ήταν σημαντικό επίσης να οριστούν στη θέα προστασίας για να αποφευχθεί κάθε μορφή ιατρικού τουρισμού αλλά να υπάρξει και αρκετή ευελιξία στο κείμενο προς όφελος της διάγνωσης από τις δύο πλευρές των συνόρων και σκέφτομαι ε, και τις σπάνιες ασθένειες και κλείνω λέγοντας ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να αγωνιστούμε για να προωθήσουμε αυτή την Ευρώπη της υγείας την οποία όλοι θέλουμε. Κύριο έχει το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Εισηγήτρια δεν υπάρχουν ιδανικά δικαιώματα, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά αυτή η οδηγία μας δίνει πολύ περισσότερες ελπίδες από ότι φόβους. Παρόλες τις αλλαγές, η Ευρώπη έχει μεγάλες διαφορές και αντιθέσεις. Ε, λόγω της σημασίας της ε, περίθαλψης υγείας εκφράζονται πολλοί φόβοι από τις φτωχές χώρες, ε, χώρες που έχουν δημοσιονομικά προβλήματα και οικονομικά, να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες ε, υγείας σε χώρες ε, υπομετάλλαξη είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ε, για τους ασθενείς από τις χώρες που ανέφερα. Ε, οι κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλη πρόκληση, αλλά η οδηγία αυτή θα πάρα, προωθήσει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και θα επισύρει την ε, προσοχή πάνω στην υποχρηματοδότηση της ε, ιατρικής περίθαλψης, όχι μόνο λόγω έλλειψης ικανοτήτων και δυνατοτήτων, διότι επειδή υπονομεύονται ε, τα βασικά αγαθά που έχουν οι λαοί της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ που θα υποστηρίξετε ε, την οδηγία ανεξάρτητα από την μορφή των προστατευτικών μέτρων που επέτρεψαν όμως το συμβιβασμό. Η ε, κυρία Γουέλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οδηγία για την κινητικότητα των ασθενών μπορεί να οδηγήσει γρήγορα να ακολουθεί και να, εξο... να υπάρξει το ελάχιστο κοινό παρονομαστή σε ό,τι αφορά την περίθαλψη των ασθενών. Δεν θέλουμε να γίνουν ασθενείς πελάτες. Η οδηγία που προτείνεται δίνει ένα εργαλείο για να χρησιμοποιούνται οι ασθενείς ως ένα εργαλείο κόστους. Δημιουργεί μεγάλη ανταγωνιστικότητα στον τομέα της περίθαλψης όταν ε, μία συγκεκριμένη θεραπεία είναι πιο φτηνή ε, κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και αποστέλλεται ο ασθενής εκεί, δεν θα χρησιμοποιείται αυτή η οδηγία. Και ο τομέας της υγείας θα υποταχθεί λοιπόν στο νεοφιλελεύθερο πνεύμα της αγοράς αντί να δώσουμε προτεραιότητα στην ευμάρεια του ασθενούς. Σας ρωτώ, λοιπόν, συνάδελφοι, θέλετε σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα να υπάρξει τουρισμός, ιατρικός τουρισμός. Πρόκειται όμως για ένα δημόσιο καθήκον του, κράτους, ε, του κοινωνικού κράτους που θα πρέπει να διατίθεται σε τοπικό επίπεδο σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κανένας ασθενής δεν θέλει δεν θέλει να βρεθεί στο εξωτερικό αν μπορεί να τύχει της ε, ίδιας ε, περίθαλψης στην οικία του. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα συστήματα υγείας, τα εθνικά συστήματα υγείας δεν πρέπει να καταστραφούν. Και πολλές φορές ο ασθενής μπορεί να τύχει καλύτερη περίθαλψη στην αλλοδαπή. Μπορεί δηλαδή να μεταβεί ο ασθενής στην Αλοδαπή όταν αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί στην ημεδαπή. Αυτό αφορά τις ιδιαίτερα σπάνιες ασθένειες μπορούμε να περιθάλψουμε και να φροντίσουμε τον ασθενή σε περίπτωση μιας σπάνιας ασθένειας. Σε μια διαφορετική χώρα θα πρέπει ο ασθενής να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μετεγκαταστήσουν τα εθνικά συστήματα υγείας. Ευχαριστώ τον κύριο Ταλή και την κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκατσισεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκροστέτ, η οποία έπρεπε να ανταποκριθεί σε μία ιδιαίτερα δυσχερή εργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ε, αποκλίσεις απόψεων στα διάφορα κράτη-μέλη το να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό μεταξύ των προσδοκιών και των δυνατοτήτων σήμερα ότι θα έπρεπε να υπάρχει και επαρκής παραγματογνωμοσύνη στο τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνεται λόγος για διασυνοριακή περίθαλψη και οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πρόσβαση σε ένα εθνικό σύστημα υγείας εκεί όπου υπάρχει επαρχή, επαρκής τεχνογνωσία. Θα πρέπει να υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα για τους ασθενείς έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα διαφορετικό σύστημα υγείας και να γίνεται και επιστροφή εξόδων. Βασιζόμαστε στα δικαιώματα των ασθενών και εξαιτίας αυτής της ε, οδηγίας θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες όχι μόνο υπέρ των ασθενών αλλά και υπέρ της βελτίωσης των συστήματων, συστημάτων υγείας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο δικαίωμα υπέρ της κινητικότητας των ασθενών και της προώθησης των δικαιωμάτων τους για να πληρωθεί αυτό το χάσμα ως προς διατάξεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ροντρίγκε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την ε, κυρία Γκροστέτ και την κυρία Ροτ ε, Μπέρεντ διότι εργάστηκαν ανελιπώς για να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία ως νομική βάση και να δώσουμε μια νέα νομική βάση έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν να επιλέγουν υπέρ της ποιοτικής περίθαλψης. Σημασία έχει ο ρόλος των κρατών μελών, ιδιαίτερα ως προς την χώρα ε, προέλευσης η οποία αναλαμβάνει τα έξοδα και τη χώρα υποδοχής. Αυτό που έχει σημασία είναι να προωθήσουμε αυτό το ποιοτικό άλμα όπως είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ γιατί θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ κρατών μελών για να μπορεί να μεταβεί οποιοδήποτε ασθενή σε οποιαδήποτε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για δικαιώματα των ε, πολιτών μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και της παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή πραγματική ισότητα, διαφορετικά τα βήματα θα είναι πολύ νοθρά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αυτή από εσά που είστε εδώ και καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θυμάστε πώς έγιναν τα πράγματα. Στην αρχή είχαμε την εισήγηση Gebhardt που θα επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφαιρέσαμε ένα μέρος και αποφασίσαμε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν ένα διαφορετικό κείμενο. Όταν αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή ε, βαθμία η ελεύθερη κυκλοφορία των υγειονομικών υπηρεσιών αφαιρέθηκε και αυτό που έμεινε είναι το δικαίωμα των ασθενών σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ θα επιζητούν ε, υπηρεσίες περίθαλψης. Θα ήθελα να τονίσω ότι καμιά φορά η ευρωπαϊκή μας ε, δέσμευση είναι κάτι περισσότερο από σημαίες και μάλλον έχει να κάνει με την ουσιαστική ελευθερία. Υπήρξαν διάφορες ανησυχίες που εκφράστηκαν από κράτη-μέλη ε, για το υψηλό κόστος κλπ. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε, αλλά είναι το σωστό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Ευχαριστώ κύριο Σνόχοτ. Εκτός μικροφώνου, ευχαριστώ. ορίζω την οδηγία αυτή που επιτέλους ε, θα εγκριθεί φαινόταν ότι είχε καταλήξει σε αδιέξοδο η νομοθετική διαδικασία και νομίζω ότι είναι επιτυχία της εισηγήτριας και της ομάδας της και φυσικά και της Βελγικής Προεδρίας που πλέον έχουμε μπροστά μας ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ικανοποιεί και το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους. Καλωσορίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα των κράτων μελών να περιορίσουν ε, την ε, γενομική περίθαλψη σε άλλες χώρες ε, γιατί στο αρχικό σχέδιο δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο και νομίζω ότι πλέον έχουμε μπροστά μας μία πρόταση όπου μπορούμε να ελέγξουμε τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε μία περίθαλψη στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό το βήμα αυτό και πιστεύω για να διατυπώσω Θεωρώ ότι ε, βοηθάμε τους 60.000 ε, ανθρώπους που βρίσκονται στα λίστες για μεταμοσχεύσεις. Ε, φυσικά έχουμε ψηφίσει σχετική νομοθεσία, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο για να περιοριστεί ο χρόνος αναμονής και έχουμε και τα εκατομμύρια ε, ανθρώπους που πάσχουν από ε, σπάνιες ασθένειες οι οποίοι πλέον μπορούν να τύχουν πιο στοχευμένης περίθαλψης ε, αν ε, την επιδιώξουν σε άλλο κράτος μέλος. Δεν πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα προκαλέσει ιατρικό τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι περιττή η ανησυχία που εκφράζει η αριστερή πλευρά του Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να μας απασχολούν τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το κείμενο είναι απότοκο μιας στεναρούς εργασίας και διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Μπάουις, Γκροστέτ και Ροτ Μπέρεντ. Έγινε μεγάλη πρόοδος διότι αυτή η νέα εκδοχή δίνει περισσότερες εγγυήσεις ως προς την ποιότητα και παροχή υπηρεσιών. Βασιστήκαμε στα άρθρα 7 και 8 και θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα. Οι περισσότεροι ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται σε χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Εκείνοι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα προσκόμματα. Γι' αυτό φοβάμαι ότι σε χώρες με ένα καθολικό σύστημα υγείας που παρέχεται σχεδόν δωρεάν, δεν θα υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις και θα δημιουργηθεί μία αγορά υγείας για τους πλούσιους. Ελπίζω όμως ε, η οδηγία αυτή να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα υγείας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και όπως και εσείς χαιρετίζω αυτή τη συζήτηση και την οδηγία και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Αλλά είμαι κάπως πιο προσεκτική, νομίζω, ότι δεν θα έπρεπε όλοι να μάθουν από εδώ ότι όλα πάνε καλά στον τομέα αυτόν. Πρέπει ακόμα να συζητήσουμε πολλά και να θέσουμε σε εφαρμογή όλα αυτά τα οποία θα ψηφίσουμε. Ε, λέχθηκε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν καθήκον να επενδύσουν στις χώρες τους για περίθλιψη ε, στους πολίτες και βλέπω ότι η Κομισιόν συμφωνεί. Καλά κατάλαβα θα πρέπει να μεταδιαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι και η χώρα μου η Ιρλανδία περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών αυτών. Θα προτιμούσαν οι ασθενείς να την περίθαλψη κοντά στον τόπο όπου κατοικούν, να έχουμε δηλαδή τοπικά νοσοκομεία και τοπικές υπηρεσίες. Η οδηγία αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά αν αναγκάσει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τις υπηρεσίες ε, στα κράτη τους και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς ε, που ε, τις χρειάζονται, διότι δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν αν χρησιμοποιούν τα δικαιώματα που τους δίνει αυτή η οδηγία οι ασθενείς. Βεβαίως, οι ασθενείς δικαιούνται να ταξιδεύουν βάσει του κανονισμού 883 για, για περίθαλψη. Δεν το γνωρίζουν, διότι αν το γνώριζαν θα είχαμε πολύ περισσότερους που θα ταξίδευαν για περίθαλψη πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες μας για αυτό το οποίο δικαιούνται. Ελπίζουμε να μην ταξιδεύουν τόσο πολύ, αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι έχουν το δικαίωμα να το πράττουν. Η κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω και εγώ την Ουγγρική Προεδρία εδώ στο Σώμα και θα ήθελα να πω καταρχήν ότι έχουμε να κάνουμε με μια οδική οδηγία Γι' αυτό έπρεπε να βγει εκτός ε, της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια του Σκιώδης και τον Τζον. Δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να αφισβητήσουμε τα κράτη-μέλη για παροχή καλής ε, περίθαλψης την οποία, την οποία οφείλουν να παρέχουν στους πολίτες τους. Εδώ μιλάμε για ποιοτική περίθαλψη για σπάνιες ασθένειες κυρίως. Επίσης μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση ορισμένων υποδομών όπως τα ιαματικά λουτρά στην Ουγγαρία που βοηθούν για συγκεκριμένες ασθένειες, αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών. Άρα μιλάμε για δικαιώματα των Ευρωπαίων και της Ευρώπης. Ο κύριος Κάζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δεδομένο ότι Πολλές φορές θεωρούμε ότι η υγεία είναι αυτονόητη όταν είμαστε υγιείς, αλλά όταν ε, αρρωσταίνουμε τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλή υγεία και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε υγειονομικά συστήματα περιθάλψης υψηλής ποιότητας, συστήματα όχι μόνο καλά και αποτελεσματικά, αλλά και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το πλεονέκτημα να έχουν πρόσβαση σε συστήματα διάφορων ε, χωρών, όπου Όποτε μια ασθένεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε κάποια χώρα. Να θυμόμαστε ότι πρέπει να είναι η τελική λύση αυτή η εναλλακτική. Η δάλος είναι πολύ ακριβή αυτή η λύση. Όπου δεν υπάρχει άλλη επιλογή θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει γραφειοκρατία και θα πρέπει να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η ασφάλεια. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τα μέσα να προστατεύουν τα εθνικά τους συστήματα από την επιβάρυνση η οποία ενδεχομένως να προκύψει από την διασυνοριακή ε, περίθαλψη. Γι' αυτό λοιπόν σημαντικό, είναι σημαντικό να υπάρχει το σύστημα της πρώτερης έγκρισης. Είναι σαφές ότι οι κανόνες που έχουμε σήμερα δεν είναι ούτε συνεκτικοί ούτε σαφείς. Έχουμε δει για παράδειγμα, και σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις, ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις για να παρέχει η Ευρώπη τις καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Σας ευχαριστώ, κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ανακούφιση το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο επιτέλου κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τα δικαιώματα των ασθενών σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή περιθαλψή για τους όρους τους οποίους ε, τόσα χρόνια του αποφάσιζε το ΔΕΚ. Χαίρομαι λοιπόν που τίθενται οι όροι για τις επιστροφές όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε πριν από 7 χρόνια για, με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω α, την κυρία Γκροστέτ και τον κύριο Μπόης που κέρδισαν τη μάχη αυτή, που κατέληξαν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό, σε μια αποδεκτή συμφωνία και θεωρώ ότι το δικαίωμα κινητικότητας θα καταστήσει πιο προσβάσιμη την περιθάλψη και θα μειώσει τους ε, χρόνους αναμονής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήτανε... Αυτό σημαίνει επίσης ότι εκπληρώνεται ένας από τους ε, βασικότερους στόχους μου σε ό,τι αφορά την περίθαλψη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Στοϊάν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την Υπουργό Γκέρι γιατί έχει, αναλάβει, έχει να αναλάβει ένα δύσκολο έργο στα πλαίσια τους ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση. Όπως ξέρετε η Ρουμανία είχε πολλές επιφυλάξεις ως προς τις προτάσεις συμβιβασμού στο επίπεδο του Συμβουλίου. Αυτές οι επιφυλάξεις δεν σημαίνει ότι αντιτιθέμεθα στη διασυνοριακή περίθαλψη. Απλώς εκφράζουμε την ανησυχία της ρουμανικής κυβέρνησης ως προς την δυνατότητα χρηματοδότησης και τη διάσταση της διασυνοριακής περίθαλψης διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα όπου οι πολίτες έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και πολύ χαμηλό ΑΕΠ. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μεταρρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι συμβαίνει στα εθνικά συστήματα υγείας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλάς. Με την κινητικότητα των ασθενών κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς μια Ευρώπη των πολιτών και η οδηγία αυτή είναι σωστή, έχει σωστές αρχές, δεν έχει μόνο ε, ένα γνωστό πατέρα, τον κύριο Μπόους, αλλά και μια γνωστή μητέρα, την κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καιρό συζητήσαμε για το σωστό τρόπο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και ξέρω ότι σήμερα ε, θέτουμε τις ε, βάσεις επί τις οποίες μπορούμε να αναπτυχθούμε. Η κατάσταση είναι περίπλοκη. Έχουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικά συστήματα και σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη αλλά και σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες η εκ των προτέρων ε, έγκριση για την περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και αυτά που ορίζονται στην οδηγία είναι σωστά για να πετύχουμε την προσωπική διασφάλιση και την προσωπική ευθύνη αλλά και αφετέρου να βοηθηθούν όλοι οι πολίτες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές που χρειάζονται. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόοδο και σε ό,τι αφορά τις σπάνιες ασθένειες, γιατί δεν είναι ε, εξοπλισμένο ανάλογα κάθε κράτος μέλος. Όλοι μπορούν πλέον να ωφεληθούν από τις ε, διατάξεις αυτές και αυτό αφορά και τους εμπειρογνώμονες για, τους, ε, για τα άτομα Τη δική μου περιοχής που βρισκόμαστε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο η οδηγία αυτή αποτελεί μεγάλο επίτευγμα και μια, έναν εμπλουτισμό σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Φερνάνδε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η παρούσα οδηγία επιτρέπει σε όλους τους ασθενείς να τύχουν περίθαλψη σε διασυνοριακό επίπεδο είναι ένα δικαίωμα που είχε αναγνωρίσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή η πρόταση διευκολύνει την πρόσβαση στη διασυνοριακή περίθαλψη ασκώντας αυτό το δικαίωμα με επιστροφή εξόδων από τη χώρα προέλευσης. Μέσα στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής οικοδόμησης και υπέρ της αλληλεγγύης βλέπουμε ότι θα έχουμε μείωση των καταλόγων αναμονής, θα υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός, καθώς και κίνητρο για τις επενδύσεις. Οι σπάνιες ασθένειες αποτελούν προτεραιότητα, θα πρέπει να γίνεται η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση. Αυτή η οδηγία ε, αποτελεί ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός για όλους τους ασθενείς. Γι' αυτό είναι παράλογο η Υπουργό Υγείας της Πορτογαλίας να αναφέρει ότι αυτή η πρόταση τάσεται υπέρ των πλέον εύπορων. Η Πορτογαλία έχει ένα ε, εξαιρετικό εθνικό σύστημα υγείας και θα ήταν παράλογο να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία για να εξυγχρονιστούμε ακόμα καλύτερα και να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές σε όσους τις χρειάζονται. Μια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εισηγήτρια την κυρία Γκροστέτ. Θα ήθελα να πω ότι αρχίζουμε με τη διαδικασία Catch the Eye. 17 ομιλητές ζήτησαν το λόγο. Επειδή είναι πολύ ε, σημαντικό αυτό το θέμα, θα δώσω το λόγο σε όλους, αλλά θα πρέπει να αρκεστείτε στο ένα λεπτό. Μετά θα σας κλείνω το μικρόφωνο. Θα ήθελα να πω προς την κυρία ε, Γκροστέτ και τον κύριο Μπόουις, προς όλους τους σκιώδους. Πιστεύω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε και πια θα αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σοκ, ένα λεπτό. Ή τα δικαιώματα των ασθενών και τα τέλος ε, στις λίστες αναμονής όλα αυτά θα τελειώσουν θα πάρουν ένα τέλος. Αυτό ακριβώς προβλέπει η οδηγία αυτή. Καταλαβαίνετε όλοι φυσικά τα προβλήματα και τις ανησυχίε χωρών που δεν μπορούν να δαπανίσουν πολλά χρήματα στην υγειονομική περίθαλψη. Κάποιοι... Κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Αν υπερψηφίσουμε την οδηγία αυτή, Ζητάμε ουσιαστικά από τα πλέον φτωχά μέλη της Ένωσης να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες. Αν καταψηφίσουμε την οδηγία θα υπονομεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών σε κάποιες από τις χώρες. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να συμφιλιώσουμε τις δύο αυτές πλευρές τα προβλήματα αυτά. Στη χώρα μου μια ε, φροντίδα στον ευωδίατρο είναι ανταγωνιστική. Ο κύριος Χάουαρτ. Με απασχολεί γιατί γίνεται λόγος για έναν ε, εθνικό ρυθμιστή ο οποίος θα πρέπει να αποφανθεί σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει την όλη ε, υπόθεση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας Γερμανός γιατρός σκότωσε τον David Gray διότι του έδωσε ένα αναλγητικό σε υπερβολικές ε, δόσεις. Υπάρχει και ο Dr. Hausman, ο οποίος ε, κατηγορείται διότι ε, φώνευσε έναν ασθενή στην Ισπανία και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαδικασία διαφοράς και παραπτώματος, παραπτωμάτων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα μέσα στα, στα πλαίσια του να μην διακυβεύεται η υγεία ασθενών από μία χώρα στην άλλη όταν μεταβαίνουν σε μία άλλη. Κύριε Μόβαιν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους της ε, Ουγγρικής Κυβέρνησης από το Συμβούλιο, δηλαδή να μας ε, πούν να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία των έξι μηνών Ουγγρικής Προεδρίας για να διαφωτίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα προβλήματα των πρώην κομμουνιστικών ε, κρατών μελών. Να τεθεί και αυτό στη συζήτηση. Όταν συζητάμε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη, πέρα από τα σύνορα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ένας ε, θεράπων ιατρός ε, εργάζεται και παίρνει μισθό 250 ευρώ. 600 ευρώ ίσως. Είμαστε σοβαροί λοιπόν. Είστε σοβαροί όταν υποβάλλετε τέτοιες προτάσεις. Δεν είναι ανήθικο να χαιρόμαστε για τη γέννηση μιας τέτοιας νομοθεσίας στην Ευρώπη. Και κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Is not here. So Ma ei arvanud, vabandage, et Δεν ε, πίστευα ότι θα μου δίνετε το λόγο τόσο γρήγορα. Ζητώ συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός ως προς την διασυνοριακή περίθαλψη. Αυτό όμως που με απασχολεί είναι ότι ακούστηκαν φόβοι για ιατρικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ανησυχούν για το, το επίπεδο ζωής που ισχύει σε ορισμένες χώρες σε σχέση με ορισμένες άλλες, διότι πολλοί ασθενείς θα προσέλθουν από φτωχότερες χώρες και θα υπάρχουν ε, μακριές λίστες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν το επιθυμούμε, διότι τα επιστρεφόμενα έξοδα θα χορηγηθούν, θα καταβληθούν ανάλογα με τα εκάστοτε ε, κρατικά δεδομένα. Η σημασία της περίθαλψης είναι γνωστή σε όλους. Υπάρχουν όμως επιπτώσεις στα εθνικά συστήματα υγείας. Υπάρχουν ανησυχητικοί τομείς τους οποίους αντιμετωπίσαμε. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια οδηγία που θα ενισχύσει τα κράτη-μέλη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή περιθάλψη έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν με βάση την ρήτρα προέγκρισης έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιες ε, περιπτώσεις θα ε, προωθήσουν. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προβούν σε συγκεκριμένες επιλογές. Έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα όπου υπάρχει μία ε, αυτονομία από πλευράς κρατών. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τον Τζον Μπόουις. Kelly. Σας ευχαριστώ πολύ που ε, μου δίνετε την ε, ευκαιρία να μιλήσω και εγώ. Θα αρκεστώ στο ένα λεπτό. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει προτεραιότητες στους ασθενείς είτε πρόκειται από φτωχά οικονομικά στρώματα ή όχι θα υπάρχει μόνο απευθυντική θηρίδα για τη γνώση και την πληροφόρηση και παράλληλα νομίζω ότι αυτή η οδηγία θα ασκήσει πίεση σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προβάλλουν ικανό επίπεδο περίθελψης για όλους τους ασθενείς. Και εν θα ήθελα να πω ότι το επίπεδο περίθαλψης είναι ύψης της σημασίας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 να επισημάνω ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να συστήσουμε εθνικά ε, σημεία επαφής ε, για να ενημερώνονται σωστά οι ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό να ε, είναι γνωστές οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις όταν δίδονται προσωρινές άδειε είναι πολύ σημαντικό ο βασικός κανόνας να είναι ότι ο ασθενής δεν πληρώνει μόνος του εκ των προτέρων τις δαπάνες και για την Ουγγαρία και για άλλους ε, είναι σημαντικό όσοι βρίσκονται στα σύνορα με τη Γερμανία ή με την ε, Σλοβακία να μην συμπίπτουν οι γλωσσικοί φραγμοί με τα σύνορα ε, χωρών. δεν πρέπει που δεν είναι να υπάρχει γλωσσικός φραγμός για να εμποδίζει τους ασθενείς ε, και να τους ε, αφαιρεί μια σωστή ε, θεραπεία διασυνοριακή θεραπεία είναι μία προϋπόθεση έτσι ώστε οι ασθενείς να την χάνουν τις βέλτιστης δυνατής ε, θεραπείας και ε, με σαφείς κανόνες ε, μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας πρέπει να δίνουμε πληροφορίες στους ασθενείς και να στηρίζουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι λοιπόν σημαντικό να διασφαλίσουμε την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τις διασυνοριακές η η ιατρική μέρημνα. Ε, οι ασθενεί πρέπει να είναι ενημερωμένοι και θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, το σύστημα που υπάρχει να την χάνουν της ελάχιστης ε, εκμετάλλευσης μέσα στους υπάρχοντες κανόνες προάγοντας ε, αποτελεσματικά συστήματα διασυνοριακής ε, θεραπείας ε, θα εφαρμόσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα οδηγία. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ομιλητές που συνέταξαν αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο. Πολλοί αντιμετωπίζουν ασάφειες ε, όσον αφορά ε, στην παροχή ε, υπηρεσιών υγείας σε άλλα κράτη-μέλη. Οι συνταγές που δημοσιεύονται σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζονται σε άλλα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα που εφαρμόζεται είναι πολύ περίπλοκο και είναι και πολύ περίπλοκο να έχει κανείς πρόσβαση στην ενημέρωση. Η επιστημονική πρόοδος δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη. Το νέο λοιπόν σύστημα επιτρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς και ενδεχομένως να επηρεάσει και θετικά το σύστημα μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Για κολλήνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η διάταξη είναι σαφώς ε, μια θετική οργάνωση και γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε την εισηγητρία και όλους ε, τους ε, άλλους που φρόντισαν για τον ορισμό και το περιεχόμενο αυτής της διάταξης. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα επιλογής στον ασθενή, ε, αυτό σε στενή συνεργασία με την ελευθερία της ε, μετακίνησης που είναι κάτι χαρακτηριστικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει η θεραπεία αυτή να προσφέρεται τόσο στις σπάνιες ασθένειες όσο και στις πολύ ειδικέ που απαιτούν μια ταχεία απάντηση η θεραπεία ε, και η άμεση θεραπεία είναι ένα δικαίωμα στην υγεία. Η υγεία πλέον γίνεται ηλεκτρονική, θεραπεύεται με ηλεκτρονικούς τρόπους και γιατί όχι. Αυτή λοιπόν η διάταξη θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει σε μια ε, πραγματική ευρωπαϊκή παροχή υπηρεσιών ε, σε πολύ ψηλό επίπεδο, τόσο τεχνολογικό όσο και από πλευράς προσωπικού. Ευχαριστώ το λόγο κυρία Σεφάλοβα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, στόχο αυτή τη συμβαστική πρόταση μετά από διετή διαπραγματεύσει είναι η εξασφάλιση τη νομική αφήνεια και τη ασφάλεια δικαίου για ασθενεί ε, με διασυνοριακέ διαστάσει ε, στη θεραπεία. Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών και υπάρχουν και τεράστιε διαφορέ μεταξύ των οικονομικών συνθήκων ε, υπό τις οποίες παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς. Στην Τσεχία έχουμε μαζικές παρετήσεις ιατρών εξαιτίας ακριβώς των περιπλοκοτήτων και των προβλημάτων που υπάρχουν. Ελπίζουμε με τη νέα πρόταση οι ασθενεί πραγματικά να αποφεληθούν από διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, αλλά χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να αποτιμήσουμε τις συνέπειες, ελπίζουμε θετικές αυτή τη οδηγία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Όμεν Ράιτεν. Αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μικολάσικ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτριά μας για την ε, προσπάθεια που έκανε σε αυτή την ε, νομοθετική πρόταση για να βελτιώσει την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής ε, περίθαλψης. Η κατάσταση μέχρι στιγμής ήταν ασαφής και αβέβαιη, κάτι που δημιούργησε τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα για τις σπάνιες νόσους. Χαίρομαι γιατί η νέα οδηγία περιλαμβάνει ειδικέ διατάξεις για τους ε, πάσχοντες από σπάνιες νόσους. Πιστεύω ότι αυτή η νομοθετική πράξη θα εξυπηρετήσει όλους τους ασθενείς, όχι μόνο αυτούς που έχουν κάποια οικονομική άνεση. Επίσης θα ευνοήσουμε την κινητικότητα των ε, ασθενών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση ε, στη διασυνορική θεραπεία στην Ευρώπη μέχρι τώρα υφίστατο κάποιους ε, περιορισμούς ε, και αυτό οφείλεται σε μακρά αναμονή, σε διαφορετικό σύστημα αποζημιώσεων και βεβαίως και στο ότι είχε και ο καθένας τη δική του ερμηνεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό, διότι θα ξεκαθαριστούν τα διοικητικά θέματα και θα είναι καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι προδιαγραφέ ποιότητα ε, τη ε, θεραπεία. Με την ε, θέσμηση των ενημερωτικών γραφείων, ο ασθενή μπορεί να ενημερώνεται για τι θεραπείε που προσφέρονται σε άλλα κράτη-μέλη και για τι διαδικασίε αποζημίωση. Αυτή λοιπόν είναι μια ευκαιρία η οποία δεν βασίζεται πλέον σε οικονομικά στοιχεία αλλά στο πραγματικό δικαίωμα επιλογής το οποίο πλέον ε, είναι ε, πολύ πιο ε, συνειδητό στους ασθενείς. Ευχαριστώ κυρία Μαρκουναϊτέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγητριά μας, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτού του πολύ σημαντικού εγγράφου. Γιατί πραγματικά ήταν χρονοβόρα διαδικασία, ήταν μακρύ το ταξίδι και καταλήξαμε στη συμβαστική λύση που δεν είναι φυσικά αποδεκτή από όλους. Υπάρχουν κάποιοι που την αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό γιατί φοβούνται μήπως εξωθήσουμε τους ασθενείς σε ένα είδος ιατρικού τουρισμού. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από πιθανή πα... κακή εφαρμογή της οδηγίας. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και να αναζητούν τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες και την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχουν όμως και γλωσσικοί φραγμοί και προβλήματα έλλειψης ενημέρωσης. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε κάποια σημεία επαφής και να βελτιώσουμε την παροχή ατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους και μόνο με εναρμονισμένη προσπάθεια θα καταλήξουμε σε αγαστά αποτελέσματα. κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Συντάμε μια οδηγία που πραγματικά λύνει το πρόβλημα χρήση υπηρεσιών υγεία σε άλλα κράτη-μέλη. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών γίνεται ήδη, όμω η οδηγία εναρμονίζει και κανονίζει, ρυθμίζει του όρου που θα γίνουν αυτή, αυτή η χρήση των υπηρεσιών. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι οι υπηρεσίε υγεία πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα και να, να τις βρίσκει ο πολίτης τοπικά, στον τόπο που, που, όπου διαμένει. Όμως υπάρχει ανάγκη πολλές φορές να προσφύγουμε και σε υπηρεσίες υγείας άλλων κρατών, ιδίως για σπάνιες ασθένειες και νέες θεραπείες. Ε, χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα και χαιρετίζω το γεγονός ότι γίνεται ειδική αναφορά στις υπηρεσίες υγείας ε, θερμών ε, πηγών και ιαματικών πηγών είναι πάρα πολύ σημαντικό. η χρήση τους επιτρέπει με λίγους πόρους να βελτιώσουμε την πρόληψη και θεραπεία πολλών ασθενειών και μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την υγεία και των ασφαλιστικών μας ταμείων. και επίτροπε σας καλώ πραγματικά να υπάρξει μια πρωτοβουλία για την προώθηση των υπηρεσιών αυτών. Το λόγο έχει η κυρία Καρβάγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κάποιους κανόνες προκειμένου να διευκολύνει την ε, πρόσβαση σε παροχή διασυνοριακών υγειονομικών ε, υπηρεσιών που θα είναι ασφαλείς και θα εξυπηρετήσουν τον ασθενή. Νομίζω ότι έτσι τηρούμε τις αρχές της οικουμενικότητας, πρόσβαση στη βιωτική υγειονομική περίθαλψη, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Είναι εμφανή τα αποτελέσματα για τους ασθενείς, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους και περίπλοκες. Γιατί οι ασθενείς αυτοί θα έχουν πια πρόσβαση σε κέντρα αριστείας, σε κορυφαίες κλινικές που ειδικεύονται στον τομέα της ε, νόσου που τους ταλανίζει. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και να συγχαρούμε το Συμβούλιο, την Επιτροπή αλλά και τη συνάδελφο Γκροστέτ για το εξαιρετικό της έργο γιατί μας βοήθησε να μετατρέψουμε σε πραγματικότητα αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ κύριε Καρβάλιο. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία του Catch the Eye με την παρέμβαση της κυρίας Αντιγόνης Παπαδοπούλου. Η υγειονομική στι μέρε μα. η παρούσα οδηγία δημιουργεί τι προποθέσει για μια ευρώπη χωρί σύνορα στον ιατρικό τομέα. οι πάσχοντε από χρόνιε σοβαρέ παθήσει μπορούν πια να απολαμβάνουν εξειδικευμένε θεραπείε να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και πληρέστερη πληροφόρηση από τα σημεία επαφή καθώ επίση μηχανισμού κάλυψη των εξόδων χωρί ταλαιπωρία. η νέα κοινοτική οδηγία δημιουργεί νέε προκλήσει πιέσει για εξυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων υγείας στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναντίλεκτα την ανάγκη για διαρκή δικτύωση και συνεργασία όλων των ιατρικών συστημάτων των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο πάντα την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την πρόθεση της ηλεκτρονικής υγείας και οπωσδήποτε τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της συνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή είναι μια πρόκληση που πρέπει να Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ολοκληρώνεται εδώ ο γύρος των συναδέλφων ε, που συμμετείχαν στη διαδικασία Κατσδιάη και θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο κύριο Τζον Ντάλι για να απαντήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διάφορες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το μέγα επίτευγμα ε, ε, κατάληξη της οδηγίας αυτής. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίνεται η οδηγία. Πρέπει να πω ότι δεν ε, συμφωνώ με την υπόνοια ότι αυτό ευνοεί τον ιατρικό τουρισμό ή βοηθάει τις ασφαλιστικές εταιρείες να μειώνουν το κόστος. Όχι. Είναι αντιθέτως διαβεβαίωση ότι καλύτερα μπορούν να τυχάνουν ιατρικών υπηρεσιών οι ασθενείς χωρίς γραφειοκρατία που πολλές φορές είναι μεγάλο εμπόδιο. Είναι πραγματικά αυτή η οδηγία καμπή για τους ασθενείς και για την ενίσχυση της Ευρώπης της υγείας θα πρέπει να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Ροτμπέρεντ και η κυρία Μαγκίνες και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι κίνητρο πλέον αυτό για τα κράτη-μέλη να επενδύσουν ε, στα συστήματα υγείας τους, διότι έχω πει και δημόσια επανειλημμένα αναφερόμενο στην οδηγία αυτή ότι δεν θέλουμε να κάνουμε ομάδε τους πολίτες μας να ταξιδεύουν, να περιφέρονται, αλλά να έχουν την καλύτερη θεραπεία που μπορούν να έχουν στις χώρες τους με την οδηγία αυτή τα δικαιώματα των ασθενών ε, κατοχυρώνονται στην νομοθεσία για τη διασυνοριακή περιθαλψή τους. Αλλά ε, το έργο μας δεν σταματά εδώ. Και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στα όσα είπε η κυρία Παρβάνοβα και ε, στην ερώτηση που έκανε για ενδεχόμενες προτάσεις που εκκρεμούν για τη διαλειτουργικότητα. Πρέπει να πω ότι η διαλειτουργικότητα είναι πραγματικά κομβική σημασία και για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και για τη συγκεκριμένη οδηγία για να γίνει λειτουργική και να μπορεί να εφαρμόζεται. Γιατί πώς αλλιώς να εφαρμοστεί με καλό τρόπο, με σωστό τρόπο αυτή η οδηγία αν δεν είναι συμβατά τα συστήματα υγείας και της ηλεκτρονικής υγείας των κρατών μελών. Ε, ε, Βεβαίω είναι πολύ σημαντική η διαλειτουργικότητα και ο συντονισμό για να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγεία τη περίθαλψη και να είναι βιώσιμη αυτή. Τώρα προσβλέπω στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να δούμε να γίνεται πραγματικότητα, να εφαρμόζεται σωστά και να υλοποιείται αυτή η οδηγία σε όλα τα κράτη της Ένωσης. Απομένουν να γίνουν πολλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό για να βεβαιωθούμε ότι η συνεργασία των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη θα γίνει πραγματικότητα. Μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα ότι θα συνεχίσω ε, αυτό το στόχο με όλη μου την ενέργεια και την αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα δώσουμε το λόγο τώρα τώρα στην κυρία Γκιορή, την οποία καλωσορίζουμε ε, ε, ε, ως εκπρόσωπο της Νέας Προεδρίας. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ στα Ισπανικά Υπουργό. Καλωσύνη σας κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Βουλευτές, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητή κυρία Συγήτρια, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πάρα πολύ ε, χρήσιμη και ωφέλιμη. Τα θέματα αυτά είναι δύσκολα και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια μας ταλαιπώρησαν ε, σε διαπραγματεύσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που οι περισσότεροι βουλευτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην οδηγία αυτή. Βεβαίως και δημιουργεί ένα καθεστώς πλέον πιο διαφανές ε, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ουγγρική Προεδρία Τη οποία το πρόγραμμα και οι προγραμματικέ δηλώσει θα συζητηθούν αύριο, ε, θέλει να εστιάζει πάντα στον άνθρωπο και στον πολίτη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Βεβαίως ε, τίποτα δεν είναι τέλειο ότι είναι ανθρώπινο ε, προϊόν. Το είπε και ο κύριος Ντάλι. Μπορούμε να βελτιώσουμε και την οδηγία αυτή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για την οδηγία για τι υπηρεσίε, για την εσωτερική αγορά και πώ αυτό εφαρμόζεται στα δικαιώματα των ασθενών. Βρέθηκε έξυπνη λύση. Θα θυμάστε τι είχε γίνει με την οδηγία για τις υπηρεσίες, τι θύελες είχε προκαλέσει. Νομίζω η παρούσα προσέγγιση είναι πολύ καλύτερη και η συζήτηση από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των ασθενών και όχι των υπηρεσιών. Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών για να φτάσουμε σε ένα στόχο ε, καλύτερης παροχής ε, υπηρεσιών υγείας στους ε, ασθενείς και στους πολίτες μας. Νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτό το στόχο. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η ελευθερία της επιλογής της περίθαψης πέρα από την ποιότητα, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη που είναι σημαντικές αρχές και θα πρέπει να πριτανεύουν. Αλλά ε, η ελευθερία της επιλογής ήταν μια επιπλέον αρχή που προσθέσαμε στον κατάλογο αυτό. Δεν είναι δικό μας επίτευγμα, είναι επίτευγμα της Βελγικής και της Ισπανικής Προεδρίας, αλλά χαίρομαι και δικό σας βεβαίως, μέλη του Κοινοβουλίου, χαίρομαι που θα δώσουμε συνέχεια, που μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση τώρα με την τοποθέτηση της κυρίας Γκροστέτ Υγητρίας για δύο λεπτά. Επ' ευκαιρία θα ήθελα, κυρία Γκροστέτ, να σας συγχαρώ για την τόσο καλή δουλειά που έκανε και εκείνη και οι σκιώδεις ηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων σε ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο, πολύ ευαίσθητο και λεπτό και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη δημοσιότητα γιατί είναι ένα από τα θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες και των 27 κρατών μελών. Έχετε το λόγο κυρία Γκροστέτ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτω με την άποψή σα. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω του πολλού ευρωβουλευτέ που μίλησαν καθ' όλη τη διάρκεια τη συζήτηση για να υποστηρίξουν την οδηγία αυτή. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω το σκιώδη εισηγητή κάθε πολιτική ομάδα Όλοι συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπω την Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Είναι πολλοί συνάδελφοι, δεν μπορώ όλου να του απαριθμίσω. Να του ευχαριστήσω, λέγω, γιατί συμμετείχαν ενεργά και επέτρεψαν στι 21 Δεκεμβρίου να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο και αύριο να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Στους συναδέλφους που εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξει για το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό μεταξύ άλλων, θα ήθελα να τους πω όχι, θα φροντίσουμε να μην ε, υπάρξει αυτό και υπάρχει ασφαλιστική ρήτρα και δικλίδα στην οδηγία. Προβλέπεται αυτό για τα κράτη-μέλη για να μπορούν να προγραμματίζουν τις υπηρεσίες υγείας τους και τις υποδομές τους και να διατηρείται αυτό. Όλα αυτά ακριβώς γίνονται για να αποφευθεί ο ιατρικός τουρισμός σε εκείνους που θεωρούν ότι η οδηγία αυτή δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, απαντώ, έχετε δίκιο. Και εγώ θα επιθυμούσα να είναι μεγαλύτερη πρόοδος, αλλά σήμερα οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι είναι τα πρώτα μόνο στάδια και βλέπω ότι ο Επίτροπος Ντάλι που μας βοηθήσε πάρα πολύ συμφωνεί μαζί μου. Θα φροντίσουμε όλοι μαζί λοιπόν να μεταφερθεί η οδηγία αυτή στα κράτη-μέλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στα επόμενα δυόμιση χρόνια θα έχει εφαρμοστεί και θα πρέπει όλοι στα κράτη-μέλη μας να επαγρυπνούμε έτσι ώστε η οδηγία αυτή να είναι υπέρ των δικαιωμάτων των ασθενών. Τελειώνοντας θα σας πω ότι αύριο η ψηφοφορία είναι αποφασιστική σημασίας. Περιμένω από εσά να έχουμε μεγάλη επιτυχία γιατί αυτή την επιτυχία θα την αφιερώσετε στους ασθενείς. Επιτέλους θα τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα σε μια ποιοτική υγεία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκροστέτ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η όλος παραδόξως κοινή συζήτηση για την όσο του Αλσχάιμερ αφενός και τους εισπνευστήρες για αφετέρου.